από τις ομάδες ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, EFDD και ENL ορισμένα αιτήματα τροποποίησης της σύνθεσης και διορισμού στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες. Οι διορισμοί αυτοί θα εμφανιστούν στα πρακτικά της τρέχουσα συνόδου. Αν δεν, αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών, οι διορισμοί αυτοί θα θεωρηθούν ότι εγκρίνονται.